Kolleginnen und Kollegen, colleagues, let's open the meeting. Συνάδελφοι, ξεκινάει η συνεδρίαση. Do you have any remarks to... Έχετε σχόλια για την ημερήσια διάταξη, παρακαλώ. Όχι. Ανακοινώσεις του Προέδρου. Νομίζω ότι θα πρέπει να ζητήσουμε από τον εισηγητή μας αύριο για το, τον εισηγητή μας για την πρώην Γεκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας να μας εξηγήσει την κατάσταση που αντιμετωπίζουμε εκεί μετά από τα όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια του Σαββατοκυριακού. Αυτό θα αποτελούσε λόγο συζήτηση και ίσως θα μπορούσαμε λοιπόν να το κανονίσουμε. Πρακτικά. Κανένα πρόβλημα? Όχι. Και τώρα λοιπόν περνάμε στο πρώτο επί της ουσίας σημείο, ανταλλαγή απόψεων με τον Τζόρτζι Μαργκελασβίλη, πρόεδρο της Γεωργίας. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε που ήρθατε εδώ και που αφιερώνετε το χρόνο να συζητήσετε σημαντικά ζητήματα μαζί μας. Είμαστε λίγο πριν από την σύνοδο της Ρήγα εταίρους και φίλους εμπεριέχει της ε, γενικότερης ε, γειτονία, σημαντικό ρόλο για όλες αυτές τις χώρες αλλά και για εμάς, θα ήθελα να τονίσω το δικαίωμα των εθνών του τμήματος αυτού του κόσμου, του τμήματος αυτού της Ευρώπης, ε, να έχουν επικυριαρχία, να λαμβάνουν τις αποφάσεις τους, το οποίο περιλαμβάνει και την ενδεχόμενη εφαρμογή συνθήκων που έχει συνάψει με την Ευρωπαϊκή Ένωση, για παράδειγμα, και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να επιδείξουμε υποστήριξη κατά τέτοιων πιέσεων. Πράξεις ε, επίθεσης από τους μεγάλους γείτονες προς την Ουκρανία αλλά και προς τη δική σας χώρα. Και η δική σας χώρα δυστυχώς έχει εμπειρία με αυτό. Και γι' αυτό λοιπόν νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να αποτελέσει τον υπαριθμό ένα σημείο στο οποίο θα πρέπει να συμβάλλουμε, συμφωνία σύνδεσης και ιδιαίτερο ελευθέρου εμπορίου προκειμένου να μπορέσουν να εφαρμοστούν σε αμφότερες τις πλευρές. Προκειμένου και οι χώρες αυτές να έχουν την δυνατότητα στη διαδικασία μετασχηματισμού που περνούν και που χρειάζονται να έχουν την ευκαιρία λοιπόν να αναπτυχθούν με σωστό τρόπο προς το κράτος δικαίου, τη δημοκρατία και κυρίως προς την κοινωνική και οικονομική τάξη που θα δώσει στους πολίτες σας ε, μια καλύτερη προπτική για τη ζωή τους. Νομίζω ότι συζητήσαμε και το θέμα της, ε, των διευκολύνσεων, της απελευθέρωσης του καθεστώς των θεωρήσεων και στην ε, συνεδρίαση των Εθνικών Κοινοβουλίων της Αντίστοιχης Επιτροπής συμφωνήσαμε ότι αν δεν υπάρχει δυνατότητα άμεσης απελευθέρωσης του το θεωρήσεων να υπάρχουν free visas ε, για τους νέους, για το καλοκαίρι, για τη Γεωργία, προκειμένου να μπορέσουν να ταξιδέψουν στην ε, Ευρώπη και στην Ουκρανία, αλλά και για τη Ρωσία. Θα ήταν πολύ πιο θα ήταν ευεργετικό να ταξιδεύουν πιο πολλοί νεαροί Ρώσοι στην Ευρώπη. Νομίζω ότι θα είχαν λιγότερε δυνατότητε να πέσουν θύματα προπαγάνδας. Θα σα δώσω λοιπόν το λόγο να συζητήσουμε τέτοια ζητήματα. Και στη συνέχεια θα δώσω το λόγο στον κύριο Καρύμ. Α, δεν έχει καταφτάσει ακόμη. Πρόεδρε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Αγαπητοί Ευρωβουλευτές, αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή που βρίσκομαι εδώ. Και ιδιαίτερα αυτή ακριβώς τη στιγμή, μια στιγμή που ετοιμαζόμαστε για ένα από τα πιο σημαντικά και ουσιώδη βήματα της εξωτερικής αλλά και της εσωτερικής μας πολιτικής, που είναι η διάσκεψη κορυφής της Ρήγας. Θα ήθελα να σας παρουσιάσω συντομία κάποιες απόψεις και σκέψεις μας για την επικείμενη διάσκεψη κορυφής, να σας πω πώς ετοιμαζόμαστε για αυτήν και ποιε είναι οι προσδοκίες μας. Το 2014 ήταν μια σημαντική χρόνια για τη Γεωργία αλλά και για την Ουκρανία και για την Ευρώπη ολόκληρη. Και ανέκτησε μερικά πολύ σοβαρά ζητήματα κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους και θα πρέπει με κάποιο τρόπο το 2015 να δώσουμε κάποιες απαντήσεις για τα ζητήματα που προέκυψαν το 2014. Ένα τμήμα των απαντήσεων, κατά τη γνώμη μου, είναι συνειφασμένο με τη διάσκεψη κορυφής της Ρήγας και των αποφάσεων που θα ληφθούν εκεί. Και επίσης ε, θα εξαρτηθεί από την απάντηση των φίλων και συμμάχων μας ε, ως προς την κατάσταση και τις περιπλοκές στην Ουκρανία, αλλά και γενικώ τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στο θέμα της πολιτικής γειτονίας. Η Γεωργία εισήλθε στην πολιτική γειτονία σε ενεργά το 2009 λίγο μετά τον πόλεμο δηλαδή, σε πολύ χαλεπούς καιρούς για την πατρίδα μου και η ανατολική εταιρική σχέση δημιούργησε, δημιούργησε για μας ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα, ένα θεματολόγιο που το χρησιμοποίησαμε δραστήρια και ενεργά την τελευταία πενταετία. Στη χώρα μου υιοθετήσαμε μια πολύ φιλόδοξη μεταρρυθμιστική ε, ατζέντα είχαμε εντατικό διάλογο με, τις, με τους εταίρους μας και χρησιμοποίησαμε την τελευταία μετα, πενταετία για να μεταρρυθμίσουμε την ε, πατρίδα μας, να την αναπτύξουμε το σύστημα αξιών μας ε, και να αναβαθμίσουμε τη χώρα εσθενιζόμενοι τους στόχους της ε, ανατολικής εταιρικής σχέσης. Και μετά την υπογραφή της Συμφωνίας Σύνδεσης διατρανώσαμε τις βλέψεις μας για την ε, ευρωπαϊκή προοπτική. Και η γεωπολιτική, ο ε, γεωπολιτικός μας προσανατολισμός αυτό δείχνει. Και δεν ήταν μόνο κυβερνητική επιλογή, αλλά και ε, επιλογή της κοινωνίας μας και της πολιτικής μας ανέκαθεν. Ετοιμαζόμαστε λοιπόν για αυτό το σημαντικό γεγονός και έχουμε κάνει πολλά. Έχουμε εκπονήσει ένα εθνικό πρόγραμμα που αντικατοπτρίζεται και στις εκθέσεις που έχουν συντάξει οι Ευρωπαίοι εταίροι μας. Οπότε προσβλέπουμε στη διάσκεψη κορυφής της Ρήγας σε ένα γεγονός που θα δείξει και θα περιγράψει με σαφήνεια τα επιτέγματα της Γεωργίας και θα δώσει μια σαφή απάντηση στα ερωτήματα που έθεσα προηγουμένως. Τα ερωτήματα είναι τα εξής. προς τις χώρες που βρίσκονται κοντά στη Ρωσία. Οι χώρες αυτές, τα έθνη αυτά, αξίζουν μια ευκαιρία να είναι ελεύθερα δημοκρατικά, να πραγματοποιούν ελεύθερα τις επιλογές τους. Αξίζουν αυτές οι χώρες στήριξης και προστασίας από τους φίλους τους. Πώς θα οικοδομήσουμε το μέλλον αυτών των δύο οικονομικών μπλοκ που ουσιαστικά χώρισαν τις έξι χώρες της Ανατολικής εταιρικής σχέσεις, Τελωνιακή Ένωση και Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου με την Ευρώπη. Στο διάλογο με τους φίλους της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης διαπιστώνουμε σαφώς ότι οι χώρες που υπέγραψαν τη συμφωνία CFTA, Ελεύθερο Εμπορίου και, όσους, και όσοι εντάσσονται στην Τελωνιακή Ένωση έχουν πολλές ευκαιρίες ε, και δεν βλέπουν φραγμούς ή αντιπαραθέσεις. Και όλα αυτά τα θέματα συνδέονται και με το μέλλον της Ευρώπης και τη σταθερότητα της Ευρώπης. Η γεωργία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για την Ευρώπη, γιατί συμβάλλει στην ενεργειακή και οικονομική της σταθερότητα, γιατί η, χώρα είναι, η Γεωργία είναι μια χώρα που συνδέει δύο πολύ σημαντικές περιοχές, της, την Κασπία και τον Εύξηνο Πόντο και είναι σημαντική χώρα διαμετακόμισης ε, πετρελαίου και φυσικού αερίου. Οπότε οι φίλοι και οι σύμμαχοί μας ε, ενδιαφέρονται για το μέλλον μας. Το ίδιο και οι γειτονικέ μας χώρες. Με όλα αυτά τα ερωτήματα κατά νου λοιπόν ετοιμαζόμαστε δραστήρια και ενεργά για τη διάσκεψη κορυφής της Ρήγας. Μάλιστα έχουμε εργαστεί πολύ σκληρά και άοκνα και πιστεύουμε ότι και μετά τη Ρήγα θα συμβάλλουμε στην ανάπτυξη της γεωργίας θα συμβάλλουμε στην ε, υλοποίηση του, των βλέψεων των ευρωπαϊκών της Γεωργίας, ώστε να καταλήξουμε στον απότερο σκοπό μας, που είναι η ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. President. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κύριε Μαμίκινς. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εξοχότητά σας. Είναι μεγάλη τιμή που σας καλωσορίζουμε εδώ στην Επιτροπή ΑΘΕΠ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και όντω. είναι μεγάλη χαρά να δούμε που βλέπουμε ότι η Συμφωνία Σύνδεση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωση και Γεωργίας, η οποία επικυρώθηκε τον προηγούμενο Δεκέμβρη, εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εφαρμόζεται. Πριν από δύο εβδομάδες ήμουν εγώ ίδιο στην Γεωργία και με μεγάλη ικανοποίηση διαπίστωσα ότι ο κόσμο στους δρόμου ήδη ωφελείται από την προσέγγιση της Γεωργίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πραγματικά σπουδαία η εμπειρία και είχα επίσης την χαρά να διαπιστώσω ότι οι μεταρρυθμίσεις συνεχίζονται και αν θα μπορούσα να προβώσω κάποια σύσταση θα πρότεινα να μην σταματήσετε γιατί οι μεταρρυθμίσεις οι οποίες έχουν εφαρμοστεί με ταχύτατους ρυθμούς, με εξαιρετικό τρόπο από πλευράς της Γεωργίας και εννοώ και την κυβέρνηση αλλά και τον λαό, τον κόσμο στη Γεωργία δεν είναι μόνο μεταρρυθμίσεις με σκοπό μόνο τη μεταρρύθμιση, αλλά αποτελούν μια επένδυση πραγματικά στις επόμενες γενιές. Σας ευχαριστούμε λοιπόν και πάλι που βρίσκεστε εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Λέω Κύριε Πρόεδρε Μαργκελεσβίλη, θα ήθελα καταρχήν να εκφράσω τη μεγάλη μου ικανοποίηση για το γεγονός ότι ήρθατε σήμερα ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων Κατά τη διάρκεια αυτής ε, της πολύ τάραχης περίοδου που διανύει η γειτονία μας ε, και είναι περισσότερο τώρα καιρός από ποτέ να δείξουμε πόσο σημαντικές είναι οι σχέσεις ε, της Γεωργίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τις δύο πλευρές επιθυμώ Μάλλον θα ελπίζω ότι η διάσκεψη κορυφής της Ρήγας δεν θα παραλείψει να τονίσει την ευκαιρία για να εμβαθυνθούν οι σχέσεις μας, να μην μείνουν όσοι έχουν σήμερα, να γίνει ένα βήμα μπροστά. Η διάσκεψη της ανατολικής εταιρικής σχέσης έχει ε, δημιουργήσει πολλές εντάσεις και συγκρούσεις γιατί η Ρωσία το αντιλαμβάνεται ως απειλή για τη δική της επιρροή. Η αντίδρασή της ήταν πολύ έντονη, αλλά το ίδιο έντονη είναι και η δέσμευση χωρών χωρών όπως η Ουκρανία, η Μολδαβία και η Γεωργία. Ενάμιση χρόνο μετά από την ε, διάσκεψη αυτή κορυφή θα ήθελα να γνωρίζω πώς γίνεται αντιληπτή η Ρωσία στην σημερινή Γεωργία. Ποια είναι η αντίληψη για τη Ρωσία στη χώρα σας. Είδα πως πρόσφατα δηλώσατε πως η Ρωσία είναι μια μεγάλη απειλή για την ασφάλεια, αλλά υπάρχει συνένεση σε επίπεδο της πολιτικής ελίτ της χώρας σας επ' αυτού. Μια άλλη ερώτηση που θα ήθελα να σας θέσω αφορά την ε, ε, εσωτερική σας πολιτική στη Γεωργία, γιατί στην ομιλία σας προς το έθνος στο Μάρτιο είπατε ότι ένα από τα σημαντικά προβλήματα της χώρας είναι συστηματικός παραλληλισμός της, νομίζω αυτό το, την φράση χρησιμοποίησατε, των ε, δομών λήψης απόφασης, που σημαίνει ότι δεν γνωρίζουμε ποιο είναι υπεύθυνο για ποιο πράγμα. Μπορείτε κάπως να μας μιλήσετε για αυτό το πράγμα, γιατί είναι πολύ ανησυχητικό, ιδιαίτερα όσον αφορά τις σχέσεις, τις θεσμικές ε, ανάμεσα στη χώρα σας και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα ήθελα να έχω περισσότερες πληροφορίες. Σας ευχαριστώ και πάλι. Ευχαριστώ. Χαίρομαι ιδιαίτερος ε, για την παρουσία του Πρόεδρου της Γεωργίας στην Επιτροπή μας, γιατί ε, ενδιαφερόμαστε ιδιαίτερα για την ανεξαρτησία της ε, Γεωργίας και μάλιστα πρόσφατα ε, εγκρίναμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισμα για την ενίσχυση της ανεξαρτησίας και της δημοκρατίας στη Γεωργία. Σίγουρα θα πρέπει να εργαστούμε όλοι και να συνεργαστούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Θα ήθελα να, μιλ... να σας ρωτήσω για την κατάσταση στις, στις κατεχόμενες βόρειες επαρχίες της Γεωργίας γιατί μας ανησύχησαν κάποιες πληροφορίες ε, για τις ε, ε, ειδικέ στρατηγικές συμφωνίες σε σχέση με τις βόρειες αυτές τις επαρχίες και την ρωσική στρατηγική παρουσία στην, στις επαρχίες αυτές. Γιατί δεν έχει αναγνωριστεί από τους υπόλοιπους αυτή η ανεξαρτησία τους. Επίσης, θα ήθελα να δω ε, πώς ε, λειτουργεί στην πράξη η αυτονομία της Αζαρίας που αυτή τη στιγμή επηρεάζεται από τη Ρωσία. Οπότε μας ενδιαφέρει ιδιαίτερη η ανεξαρτησία της Γεωργίας και φυσικά η ε, αρμονική περαιτέρω ανάπτυξη της ε, γεωργιανής δημοκρατίας. Γιατί τους τελευταίους μήνες πολύ συχνά ακούσαμε για την επιλεκτική δικαιοσύνη, για τις τεταμένες σχέσεις κυβέρνησης και αντιπολίτευσης ε, για τις ε, σχέσεις με τον ε, απερχόμενο πρόεδρο και το κόμμα του, το Ενωμένο Εθνικό Κίνημα. Πάντως σας διαβεβαιώ ότι όλοι ενδιαφερόμαστε για αρμονικές και εύρυθμες σχέσεις μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Γιατί αυτές οι αρμονικές σχέσεις αποτελούν σημαντικό, στοιχείο, σημαντικό και αναπόσπαστο στοιχείο και της δημοκρατίας αλλά και της εσωτερικής ασφάλειας οποιοδήποτε χώρας και έτσι δεν δημιουργείται και πρόσφορο έδαφος για εξωτερικές παρεμβάσεις αν εξασφαλιστεί αυτή η αρμονία. Thank you, Mr. President. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και οι φιλελεύθεροι καλωσορίζουν για τον Πρόεδρο της Γεωργίας που εκπροσωπεί ε, μία από τις πιο πλούσιες χώρες του κόσμου και έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε τις ε, δικές σας αποφάσεις. Ε. Και Άλλες χώρες ε, έχουν υποστεί κατοχή από τη Ρωσία, όπως η Μολδαβία και η Ουκρανία. Οραματίζεστε σε πιο στενή συνεργασία με τις χώρες αυτές που επηρεάζονται άμεσα από τις ε, ρωσικές παρεμβάσεις και πώς θα δημορφωθεί μια τέτοια συνεργασία. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος, και θα ήθελα εδώ πέρα να κλείσω τον κατάλογο μιλετών, γιατί θα πρέπει να ξεκινήσουμε 4 παραδάρτο με τις ψηφοφορίες. Το λόγο λοιπόν τώρα έχει η κυρία Άουταλα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, είχα ήδη την ευκαιρία να θέσω κάποιες ερωτήσεις στο ε, πρόσωπό σας αυτό το ενδιαφέρον σεμινάριο το οποίο διοργανώσατε λίγο πιο πριν ε, εδώ στο Κοινοβούλιο. Νομίζω όμως ότι θα άξιζε να αναπτύξετε λίγο παραπάνω το εξής ε, θέμα εδώ στην Επιτροπή μας. Ποια είναι η αποψή σας για τη μεταρρύθμιση του δικαστικού σώματος, γιατί όπως ξέρετε αποτέλεσε αυτό μια ιδιαίτερη ανησυχία του Κοινοβουλίου. Σε διάφορους βαθμούς μας έχει απασχολήσει το θέμα αυτό και ένα άλλο θέμα θα ήθελα να αναφέρω. Αναφέρετε την δυνατότητα να εξευρεθούν λύσεις κατά κάποιο τρόπο μεταξύ των δύο ανταγωνιστικών εμπορικών συστημάτων τα οποία έχουμε σήμερα από την άλλη, έχουμε και την ελεύθερη ζώνη εμπορίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία θα συνδεθούν πλέον και εσείς και η Ουκρανία και η Μολδαβία. Και ύστερα υπάρχει και η CIS, ε, ζώνη ελεύθερου εμπορίου Ευρασίας. Πιστεύετε ότι υπάρχει κάποιος τρόπος να απαλληλθούν οι τρομακτικές ε, πολιτικές εντάσεις που υπάρχουν λόγω της ε, ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία σήμερα και να προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε τα δύο αυτά εμπορικά συστήματα. Δεν μιλάω για πιο ήπιες κυρώσεις από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά την κρίση της Ουκρανίας. Εκτός μικροφώνου, Πρόεδρος. Thank you, Chair. Σας ευχαριστώ, αξιότιμη κύριε Πρόεδρε. Η κατάσταση ε, έχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία χρόνια και φάνηκε και στην έκθεση Πάσκου του, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και είχαμε μια μεγαλύτερη θετική ολοκλήρωση αρχικά των βαλτικών χωρών, των χωρών της Βαλτικής, αλλά και των υπολείπων. Πιστεύετε ότι η μεγαλύτερη ακόμη στρατηγική ολοκλήρωση και στη δική σου περιοχή του Καυκάσου θα ήταν δυνατή. Για παράδειγμα, με τη δημιουργία ενό τάγματο που, στο οποίο θα συμμετέχουν Γεωργία, Ουκρανία και Μολδαβία. Ευχαριστώ. Η κυρία Φωτίγκα, ευχαριστώ. Καλώς ήρθατε εξοχότατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και χαίρομαι ε, για την ευκαιρία που έχουμε να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο της Γεωργίας ε, με τον άνθρωπο που έχει, κατέχει το ύπατο πολιτικό αξίωμα στη χώρα αυτή και μάλιστα λίγο πριν το, τη διάσκεψη κορυφής της Ρήγας. Είστε μία από τις χώρες που ανέκτησαν την ανεξαρτησία τους μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης και φυσικά αξίζεται και ανεξαρτησίας και σταθερότητας και ειρηνικής ανάπτυξης. Ε, είναι αυτονόητο ότι όλες αυτές οι χώρες αξίζουν τέτοια ανεξαρτησία, ανάπτυξη οικονομική και σταθερότητα. Και αυτό θα πρέπει να είναι το μήνυμά μας στη Ρήγα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι προσιλωμένη σε αυτό το σκοπό και διατρανώνει το μήνυμα αυτό. Επίσης, θα ήθελα να σας εκφράσω τις ανησυχίες μου για την πατρίδα σας. Γιατί ήμουν ανέκαθεν πιστός και προσιλωμένος φίλος ε, στην πατρίδα σας και στην πρόσφατη μου επίσκεψη συναντήθηκα με ε, φυλακισμένους ε, πρώην πολιτικούς σας αντιπάλους μέλη του κόμματος του κυρίου Σακασβίλη και συναντήθηκα και με δικηγόρους. Ποιες είναι οι σκέψεις ως προς την προοπτική μεταρρύθμισης του δικαστικού συστήματος, ώστε να αντιμετωπιστεί αυτή η συζητήσιμη μέθοδος της ε, κράτησης, ε, της προσωρινής κράτησης και μάλιστα πριν τη διεξαγωγή δίκης. Πιστεύετε ότι και εν ώψη της διάσκεψης κορυφής της Ρήγας θα έχουμε κάποιες θετικές εξελίξεις ε, και στη δικαστική μεταρρύθμιση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν και εμείς ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Καμποτζόμπα, όπως λέτε και εσείς ε, στη Γεωργία, στις Βρυξέλλες, στην προκειμένη περίπτωση. σου αναφερθήκατε στην ευρωπαϊκή προοπτική που είναι σημαντική για την Γεωργία και για το λαό της Γεωργίας η οποία είναι βαθιά ριζωμένη στην ενοτροπία του κόσμου στην γεωργία και όταν συναντιόμαστε με ανθρώπους στη γεωργία είναι σαφές προς τα ποια κατεύθυνση θέλουν να κινηθούν οι άνθρωποι στη γεωργία προς τα που είναι προσκύμενοι για ένα πιο λαμπρό μέλλον. Σε ό,τι αφορά την περιφερειακή συνεργασία, γιατί στο Νότιο Κάφκασο υπάρχουν χώρε διαφορετικού προσανατολισμού για διάφορου λόγου, κατά πάσα πιθανότητα. Και υπάρχει ένα μεγάλο παιχνίδι γεωπολιτικό το οποίο διεξαγάγεται στην περιοχή αυτή. Αναρωτιέμαι λοιπόν το πώς έχει, λαμβάνοντας υπόψη και πώς έχει η κατάσταση ε, στην περιοχή. Τι γίνεται με την ενεργειακή συνεργασία και με τα σχετικά έργα που θα πρέπει να κατασκευαστούν στην περιοχή για να συνδεθεί καλύτερα ο Νότιος Κάφκασος με την Τουρκία αλλά και άλλες χώρες. Ποιες είναι θεωρείτε οι προοπτικές για αυτά τα τεράστια project, τεράστια αυτά έργα. E- και έτσι λοιπόν ε, έχει ένα λεπτό τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου οι βουλευτέ. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομο. Θα ήθελα καταρχήν να σα πω ότι ειλικρινά θα μπαίνω στο πειρασμό να απαντήσω διεξοδικά σε όλε τι ερωτήσει γιατί είναι πολύ ενδιαφέρουσε και σημαντικέ και μπορούν να μας διαφωτίσουν για όλα αυτά τα σημαντικά θέματα που θίξαμε. Σε ό,τι αφορά τη Ρωσία. Σχέση με τη Ρωσία. Βέβαια, η Ρωσία ήταν απειλή στην ασφάλεια της Γεωργίας και στην εδαφική ακεραιότητα και την κυριαρχία της Γεωργίας. Και αυτό δεν συνέβη μόνο το 2008. Έλεγα στους συναδέλφους ότι και στη δεκαετία του 90 είχαμε δει και στη Γεωργία κάτι που βλέπουμε σήμερα στην Ουκρανία, αυτό τον υβριδικό πόλεμο, δηλαδή κατοχή εδαφών. Και οι πρόσφατες συμφωνίες ε, με τα εδάφη αυτά της, ε, του Βορρά είναι ένα ακόμη βήμα προς την προσάρτηση. Το είδαμε στη δεκαετία του 90, στις αρχές της δεκαετίας του 90, στο τέλη της δεκαετίας του 90, το 2008 και σίγουρα η Ρωσία συνιστά απειλή. Και αυτό που συνέβη στην Ουκρανία το είχαμε βιώσει και εμείς προηγουμένως ε, στη Γεωργία. Και μάλιστα έξι χρόνια πριν. Και αυτό επαναλαμβάνεται τώρα με την Ουκρανία η Ρωσία δεν έχει ακόμη καταβάλει το τίμημα για αυτά που έκανε το 2008. Και έτσι μπόρεσε να είναι πολύ πιο γρήγορη και πιο εύκολη στις επεμβάσεις της το 2014 στην Ουκρανία. Υπάρχει αυτή η αίσθηση του, της ανασφάλειας. Ναι, υπάρχει και φυσικά αυτό που περιμένουμε είναι ένα ξεκάθαρο και χειρό μήνυμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα θέματα αυτά. Η γεωργία αξίζει ένα σαφές, ένα καθαρό μήνυμα για το δικαίωμά της να τύχει προστασίας στην ελεύθερη επιλογή της να αποτελέσει τμήμα της δυτικής κοινωνίας. Νομίζω ότι αυτή η φωνή θα πρέπει να ακουστεί πολύ πιο ηχηρά, πολύ πιο ξεκάθαρα και το ίδιο ρητά και κατηγορηματικά με τον τρόπο που μιλούν οι Ρώσοι. Γιατί ήταν σαφέ το μήνυμα τη Ρωσία. Είπαν ότι οι χώρε τη πρώη Σοβιετική Ένωση ε, βρίσκονται στη σφαίρα επιρροή του και έχουν το δικαίωμα να αποφασίζουν για αυτέ και με τη χρήση στρατιωτικών μέσων. Οπότε κάθε ε, μία από τι χώρε αυτέ. Ε, ζει υπό απειλή και για οποιοδήποτε λάθος, οποιαδήποτε αστοχία ή αβεβαιότητα θα εμφανιστεί η Ρωσία με στρατιωτικά μέσα για να επιλύσει την κατάσταση και να επιβάλλει τις αποφάσεις της. Και να συνδέσω αυτό το θέμα με το ζήτημα της ε, Τελωνιακής Ένωσης. Ε, σε σχέση με τη Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποια θα ήταν η, λύση. Σας είπα ότι όταν συζητούμε με τους ε, Αρμένιους και, τους, και λέμε ότι εκεί είναι ε, στην Τελωνιακή Συμφωνία με την ΚΑΚ και εμείς στην Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών και όταν μιλούμε με τους Λευκορώσους Θεωρούμε ότι όλες αυτές οι συμφωνίες δημιουργούν ευκαιρίες για περαιτέρω ευημερία και δεν δημιουργούν διαχωριστικές γραμμές και αντιπαράθεση. Εμείς αναζητούμε ευκαιρίες εμβάθυνση των οικονομικών σχέσεων. Ποιος όμως προσπαθεί να δημιουργήσει αντιπαράθεση και μεταφέρει τα εμπορικά θέματα σε γεωπολιτικό επίπεδο και σε θέματα υπαρξιακής επιλογής, η Ρωσία πάνω απ' όλα. Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς απέναντι σε αυτή την συμπεριφορά. Μπορούμε να έχουμε μια σαφή και ξεκαθαρή απάντηση, ένα πρόγραμμα ευρωπαϊκό για να δώσουμε σαφείς και ξεκάθαρους προσανατολισμούς για το μέλλον. Θέλουμε να δημιουργήσουμε, να πραγματοποιήσουμε μικρά και σαφή βήματα. Όχι πολιτική της αντιπαράθεσης, άσχετα με την Ουκρανία, τη Γεωργία και τη Μολδαβία. Θέλουμε να δείξουμε στη Ρωσία, να δείξουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στη Γεωργία και σε άλλες χώρες ανατολικής εταιρικής σχέσης ότι ο τρόπος σκέψης της αντιπαράθεσης μπορεί να αντιμετωπιστεί με ένα θετικό μήνυμα, με μια θετική δυναμική, με τη δημιουργία νέων ευκαιριών με τις χώρες ανατολικής εταιρικής σχέσης. για την εταιρική σχέση Γεωργίας, Ουκρανίας και Μολδαβίας. Σίγουρα αυτές οι τρεις χώρες ε, έχουν προωθήσει περαιτέρω τις σχέσεις τους μέσω της ανατολικής εταιρικής σχέσης και τις έχουν ευαθύνει υπογράφοντας και συμφωνία σύνδεση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν υπάρχει τώρα δυνατότητα περαιτέρω ε, συνεργασίας, έχουμε εταιρική σχέση σε πολιτικό επίπεδο Έχουμε υποστηρίξει αμέριστα και ρητά την Ουκρανία που υπόκειται σε εντάσεις και αντιμετωπίζει σημαντική απειλή. Και αυτό το εκδηλώσαμε σε κάθε επίπεδο. Ο Υπουργός Εξωτερικών μας ε, δραστηριοποιείται και καλεί και τους Υπουργούς Εξωτερικών αυτών των χωρών για να έχουμε ενιαίο διάλογο και ενοποιημένο μήνυμα, τουλάχιστον για τις τρεις αυτές χώρες. Οι ενώσεις, κατά τη γνώμη μου, γίνονται με βάση τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που έχει κάθε χώρα. Εμείς προσπαθούμε να αναπτύξουμε τις σχέσεις μας και να τις προωθήσουμε στο σωστό πλαίσιο με βάση το σύστημα αξιών μας, με βάση την κοινή μας προσέγγιση για το μέλλον και για την εξωτερική μας πολιτική και για τις κοινέ μας αξίες, για τα ανθρωπιστικά θέματα. Σε ό,τι αφορά την στρατιωτική συνεργασία, νομίζω ότι η απόψη στρατιωτικής συνεργασίας καλύτερα για τη Γεωργία να μπει στο ΝΑΤΟ και να αξιοποιήσει το ανταγωνιστικό πλονέκτημα του ΝΑΤΟ. Και μάλιστα αυτός είναι ο στόχος μας, η ένταξη στο ΝΑΤΟ και θα ήταν πολύ πιο κατάλληλη απάντηση για όλες αυτές τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε στην περιοχή. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις εσωτερικές υποθέσεις και τις εσωτερικές πολιτικές, είπα σήμερα ότι πιστεύω και είμαι υπερήφανος για τις μεταρρυθμίσεις που έχουν εφαρμοστεί την τελευταία διετία. Η δικαστική εξουσία ήταν από αυτές που είχαν αμεληθεί σχετικά στο δημοκρατικό μας σύστημα. Καταβάλαμε τεράστιες προσπάθειες για τη μεταρρύθμιση της. Αυτά φυσικά δεν μπορούν να γίνουν εν μία νυχτή. Είναι μια χρονοβόρα διαδικασία, περίπλοκη, αλλά την τελευταία διετία πραγματοποιήσαμε σημαντική πρόοδο. Συμφωνήσαμε και αρχίσαμε τη μεταρρύθμιση στην εισαγγελική αρχή, στο γραφείο του εισαγγελέα που είναι από τους πιο δύσκολους τομείς που καλούμαστε να μεταρρυθμίσουμε. Το γραφείο του Εισαγγελέα, η Εισαγγελική Αρχή είναι ένα τμήμα της δικαστικής, του δικαστικού συστήματος που χρήζει διεξοδικής μεταρρύθμισης. Επίσης, μεταρρύθμιση στο σύστημα των δικαστηρίων. Θέλουμε ένα σύστημα εύρυθμο, γιατί μέχρι στιγμής τα δικαστήρια δεν συνεργάζονται εύρυθμα με την εισαγγελία, κάτι που δημιουργεί πρόσκομα στην εύρυθμη απονομή της δικαιοσύνης. Επίσης, ένα θέμα που συνδέεται άμεσα με τις εξουσίες του Πρόεδρου και μάλιστα χαίρομαι γιατί το καταφέραμε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, διορίσαμε έναν υπερκομματικό πρόεδρο του δικαστηρίου και δικαστές που δεν είναι πολιτικοποιημένοι, δεν, είναι πολιτικ... δεν στηρίζονται από κανένα πολιτικό κόμμα και συνεχίζουμε αυτή την αποπολιτικοποίηση του δικαστικού συστήματος. Σίγουρα υπάρχουν κάποιες αδυναμίες και βελτιώσεις που χρειάζεται να γίνουν. Σε ό,τι αφορά το, το χρόνο κράτησης πριν τη δίκη, είναι ένα από τα επίμαχα σημεία. Δεν θέλω τώρα εδώ να επισέλθω σε συγκεκριμένες υποθέσεις και πιο αναλυτική παρουσίαση, αλλά θέλουμε να φτάσουμε στις ευρωπαϊκές προδιαγραφές, όπου ε, άνθρωποι κανονικά που δεν έχουν διαπράξει σοβαρά εγκλήματα δεν πρέπει να φυλαγγίζονται πριν την εξαγωγή της τους ή να μην φυλαγγίζονται άνω του διμήνου που είναι το ευρωπαϊκό όριο για την προσωρινή κράτηση. Πάντως σας διαβεβαιώ ότι μέχρι στιγμής ε, οι μεταρρυθμίσεις ε, έχουν εφαρμοστεί και έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο. Δεν ξέρω αν παρέλειψα κάτι. Για τις συνθήκες, ε, σας είπα τις συνθήκες, έχουμε υπογράψει και τις συμβάσεις. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εταίρους ε, και φίλους μας που αναφέρθηκαν στα σημεία αυτά και μας στήριξαν ενεργά. Σε ό,τι αφορά τη συνθήκη που υπέγραψε η Ρωσική Ομοσπονδία με την Απχαζία, το μήνυμά μας ήταν ξεκάθαρο. Σε ό,τι αφορά τη συνθήκη με την ε, Νότια Οσετία, ευχαριστούμε τους φίλους και τέρους για την κατηγορηματική του συμπεριφορά και το χειρό μήνυμα που ε, έστειλαν και πριν την υπογραφή μάλιστα της σχετικής συνθήκης από τη Ρωσική Ομοσπονδία με την Νότια Οσετία. Είπατε ότι καταστρατηγεί η συνθήκη αυτή τις διεθνείς προδιαγραφές και σας ευχαριστούμε θερμά για την υποστήριξή σας. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, για τις παρατηρήσεις σας. Θα ήθελα να δηλώσω ότι μπορείτε να εμπιστεύεστε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είμαστε με στο πλευρό σας, όπως νομίζω έχουμε αποδείξει εδώ και αρκετά χρόνια. και ελπίζω πως θα μπορέσετε να αναπτύξετε τη χώρα σας με τέτοιο τρόπο, ώστε η Συμφωνία Σύνδεσης και η Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου να μπορέσει να εφαρμοστεί πλήρως έτσι ώστε να αναπτυχθούν όλες οι προοπτικές της χώρας σας. Ελπίζουμε λοιπόν και ότι η διάσκεψη κορυφή της Ρήγα θα είναι επιτυχής. Σας ευχαριστώ πολύ.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 Κυρίε not now. Ladies and gentlemen. Κυρίες και κύριοι, Ρωσία τώρα. Ο κύριος Λανσπέρκης δεν ξέρω αν έχει κάτι να πει. Να ευχαριστήσω εκ νέου όλους όσοι συμμετείχαν στη διαδικασία προετοιμασίας του εγγράφου. Να προσέχετε, να προσέχετε, λέει ο Πρόεδρος. Μετά, μετά, περιμένετε την ψηφορία και μετά ευχαριστείτε. Αυτά. <laughs> Wir beginnen να ξεκινήσουμε λοιπόν. Τροπολογία 1. Του εισηγητή. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Σόλτς. Η ε, 165. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Και έτσι λοιπόν περνάμε στην Συμβιβαστική 2. Λίγο διαφορετική η σύνθεση αυτή τη φορά και η παρουσίαση. Συμβαστική 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και έτσι περνάμε στη συμβαστική 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και έτσι φτάσαμε στην 2.36. Μία μία προσθήκη. Ποιος είναι υπέρ της 2.36. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. Ζητείτε έλεγχος. Πέρας ψηφορίας. 26 υπέρ, 28 κατά, 2 αποχές απορρίπτεται. Doesn't help Σας βοηθάει. Άλλη μια ψήφο υπέρ, αλλά και πάλι δεν αρκεί, λέει ο Πρόεδρος. Και έτσι περνάμε λοιπόν στην ε, τροπολογία υπαριθμών 258. Υπέρ. 258. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 261. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Πώς είπατε, θέλετε έλεγχο. Θα μου κεράσετε, άμα έχω δίκιο. Ένταξη ψηφοφορία. 261. Πέρας ψηφοφορίας. 21 υπέρ, 34 κατά. Απορρίπτεται. Και τώρα περνάμε στη συμβαστική 6 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 294 υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. 296 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Στην 303. Υπέρ. Υπέρ 303. Κατά. Άποχες απορρίπτεται. Εξακολουθεί να απορρίπτεται, λέει ο πρόεδρος. Συμβαστική 8. Α, συγγνώμη, 304. Η 304 υπέρ. Κατά. Άποχες απορρίπτεται. Σεμιβαστική 8 υπέρ. Κατά άποχες εγκρίνεται. 314 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 22 Υπέρ. Κατά. Αποχές έλεγχος. Abstimmung ist geschlossen. Πέρας 22 υπέρ, 39 κατά, απορρίπτεται. 300. Η συμβαστική 9. Η, η 323. 323. Υπέρ. Υπέρ. 323. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές έγκρινεται. 3.46. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβαστική 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. Συμβαστική 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 3.49. Η 363. Η 363. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. 379. 379. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 12 υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Η 3, 94 ε, ε, υπέρ. Κατά. Τι λέτε λέει ο πρόεδρος. Η 34 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 13 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 14 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 409 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος για την 409. Die Abstimmung ist geschlossen. Πέρας ψηφορίας. Πάντα το ήξερα ότι έχει Μεγάλη επιρροή ο Σάρις Βόλσκι Απορρίπτεται. Με μία ψήφο διαφορά. Α, εγκρίνεται. Τότε ψήφισε λάθος. Όχι εγκρίνεται λοιπόν, λέει ο Πρόεδρος. Εγκρίνεται. Εγκρίνεται. 411 Σε τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Dann Abstimmung ist geschlossen. Εγκρίνεται. Και περνάμε στο δεύτερο τμήμα τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ο κύριος Χάουιτ δεν έχετε χρόνο για κυβερνητικούς ε, κυβερνητικές διαπραγματεύσεις. Καθυστερήσατε. Συμβαστική 15. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Συμβαστική 16. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. 462. Τροπολογία 462. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 463. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 17. Υπέρ. Κατά. Α, εγκρίνεται. Συμβαστική 18. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 27. Τροπολογία 27. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 19. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 20. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 21 υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. 31 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 22. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 67. Τροπολογία 67. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 23. Υπέρ. Κατά. Αποχές έγκρινεται. Συμβιβαστική. 24. Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος παρακαλώ. Mal τη stimmt Abstimmung ist geschlossen. 40 υπέρ, 26 κατά έγκρινεται. Η 79 ως προσθήκη υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 25. Η συμβαστική 25. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Έγκρινεται. 103. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. 26. 26. Συμβαστική 26. Συμβαστική 26. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 27. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 29, 28 διορθώνει ο πρόεδρο. Συμβαστική 28 υπέρ. Κατά. Αποχέ έγκρινεται. Συμβαστική 29 υπέρ. Κατά. Αποχέ έγκρινεται. Συμβαστική 31 υπέρ. Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχέ έγκρινεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Έλεγχο παρακαλώ. Der Antrag ist geschlossen. Äh, der, die Abstimmung ist geschlossen. 40 υπέρ 24 κατά μία εποχή εγκρίνεται. Και τώρα περνάμε στην 140, τροπολογία 140. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 30 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 32 Συμβαστική υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 154. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται, νομίζω. Η 154. Πέρας ψηφοφορίας. 38 υπέρ, 27 κατά εγκρίνεται. 161 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 1 και 2 υπέρ. Έχετε εδώ πέρα και έναν συντάκτη. Σε συντάκτη κυρία Σάριος Βόλσκη. Υπέρ. Κατά. Έλεγχος. Die Abstimmung ist geschlossen. Πέρασε. 38 υπέρ, 28 κατά, εγκρίνεται. Η 3 υπέρ. Κατά. Αποχές, απορρίπτεται. 4 υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. 5 υπέρ. Η 5 υπέρ. Κατά. Αποχές, απορρίπτεται. 6 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 7 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ηλεκτρονική ψηφοφορία για το σύνολο του κειμένου. Die Abstimmung ist geschlossen. Εγκρίνεται 53 ψήφοι υπέρ, 10 ψήφοι κατά 3 αποχές. Καλ... Συγχαρητήρια κύριε Λαντσπέργης. Αλλά συγχαρητήρια και σε όλους όσοι με μεγάλη σοβαρότητα προσπάθησαν να πετύχουν συμβιβασμού την τελευταία εβδομάδα, τις τελευταίες εβδομάδες μάλλον. Και τώρα λοιπόν περνάμε στην έκθεση για την Τουρκία. δικαστικό? Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μου επέστησε την προσοχή σε ένα λάθος στον κατάλογο ψηφοφορίας του ΕΛΚ. Όντως ε, είναι λάθος και σας παρακαλώ συναδελφοί να το διορθώσετε στη σελίδα 34 στην 415 ε, όπου υπάρχει αρνητικό πρόσημο, θέλουμε να μπει θετικό πρόσημο για τη συμβαστική 22 για να προσθεθεί το values αξίες δηλαδή επί των οποίων έχει ιδρυθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ παρακαλώ να μπει θετικό πρόσημο στο κατάλογο ψηφοφορίας. E Στο κατάλογο ψηφοφορία του ΕΛΚ. Δεν έχω λοιπόν κανένα σχόλιο να κάνω. Ο Πρόεδρος. Το ΕΛΚ δεν έχει και φαξ. Και άρα αναγκαστικά καταφεύγει σε αυτές τις λύσεις. Η 48. 48 υπέρ. Κατά αποχές έγκρινεται. Ας ελέγξουμε. Καλά αρχίζουμε. Πέρας ψηφοφορίας. 37 υπέρ, 29 κατά, εγκρίνεται. Συμβαστική 1 υπέρ. Κατά, α, εγκρίνεται. Η 58, 59 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται Απορρίπτεται. 61 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 2 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 74 υπέρ. 74 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Και έτσι περνάμε. Την 83. 83. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Έλεγχος παρακαλώ. Abstimmung ist geschlossen. Πέρας ψηφοφορίας. 26 υπέρ, 34 κατά, 6 εποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 3 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 91 υπέρ. Ναι, είναι 91. 99. 99. Υπέρ του Γκούναρ Χοκμάρκ. Λοιπόν, ποιο είναι υπέρ τη 99. Κατά. Αποχές. Δεν είναι βέβαιο το αποτέλεσμα. Ας ελέγξουμε παρακαλώ. 32 υπέρ, 33 κατά, απορρίπτεται. Συμβαστική 4. Υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. 107. Για 107 όσο έχει υπέρ. Κατά. Απορρίδετα. Εκατόν έντεκα. Εκατόν έντεκα, υπέρ. Κατά. Έλεγχος. Τα άψιμο είναι κλεισμένο. Περάσει. 32 υπέρ, 34 κατά απορρίπτεται. 113 ε, υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 5 υπέρ. Κατά. Αποχές έγκρινεται. Συμβαστική 6 υπέρ. Κατά. Αποχές έγκρινεται. Συμβαστική 7 υπέρ. Κατά. Αποχές έγκρινεται. 130 Τροπολογία 130 υπέρ. Κατά. Άποχες. Έλεγχος. Abstimmung Πέρας. 27 υπέρ, 32 κατά απορρίπτεται. Συμβάσει και 8 τώρα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 140 τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 139 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 141 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τι έκπληξη. Συμβιβαστική 9 υπέρ α, 148. Deutlich machen, ich kann das doch nicht auswendig lernen. Wir müssen vor 148. We have to change. Πρέπει να ψηφίσουμε λοιπόν την 148 επειδή δεν εγκρίθηκε η 140 ή 148 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική εννέα, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική δέκα, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 165 τώρα. Κάτι δεν πάει καλά όμως εδώ. Darf ich so reinschauen und mich dahin jagen? Ist doch die Liste falsch. Wir kommen 170. Στην 170 λοιπόν περνάμε. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Wir 172 υπέρ. 170 έλεγχος. Abstimmung ist geschlossen. ψηφοφορίας. 47 υπέρ, 18 κατά. Εκατόν εβδομήντα λέει ο πρόεδρος. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 173 υπέρ. Κατά αποχές έλεγχος. Η Abstimmung geschlossen. Πέρας ψηφοφορίας. 36 υπέρ, 23 κατά εγκρίνεται. 174 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 177 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 175 υπέρ. Κατά. Αποχές έγκρινεται. 175 παρακαλώ πάλι. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 176 υπέρ. Κατά. Αποχές έγκρινεται. 178. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. 179, 180, 181. Υπέρ. Κατά. Έλεγχος παρακαλώ. Πέρας. 43 υπέρ, 23 κατά εγκρίνεται. Συμβιβαστική 11 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η συμβαστική 12 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 196 εδώ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Νομίζω όμως ότι εγκρίνεται. Πέρας. 41 ψήφοι υπέρ, 22 κατά εγκρίνεται. Συμβαστική 13 υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 14 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 124. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έγκρινεται. Για την 224. Είναι δυνατόν να είναι κανείς σε κατά τροπολογία της Ρεβέκας. Περάσε. 39 υπέρ, 24 κατά. Εγκρίνεται. Οι τρεις ταυτόσημες. Τώρα. Υπέρ. Κατά. Έλεγχος. Abstimmung ist geschlossen. Πέρας. Και διάβασα τι τροπολογίε, λέει ο Πρόεδρο. Ιδιαίτερω αυτέ. 32 υπέρ, 32 κατά διακόσια είκοσι 28-229 υπέρ υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η 230 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 231 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 233 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 234 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Και αυτό θα πρέπει να με κεράσει. Die Abstimmung ist nahezu geschlossen. Σχεδόν ε, ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία. Πέρας. 20 υπέρ, 33 κατά. 235 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 236 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Kompromiss 15. Συμβαστική 15. Α, όχι, ψηφοφορία. 29 κατά, υπέρ, 31 κατά. Απορρίπτεται. Συμβαστική 15. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 16. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 17. Υπέρ. Κατά αποχές Εγκρίνεται. 263 υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. Έλαχος. Δεν ήθελα να πιω και τόσο πολλά σήμερα. Θα με κεράσετε πολύ. Άψιμος Πέρα τις Α, εδώ θα χρειαστεί να επιστρέψω το κέρασμα. Εγκρίνεται. «271, 272, υπέρ». Κατά. Αποχές έγκρινεται. 273. Ε, Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 18 υπέρ. Κατά. Άποχες. Έγκρινεται. 282. Καταπίπτει. Λάθος. 284. Υπέρ. Κατά. Ε, αποχές. Απορρίπτεται. 287. Υπέρ. Κατά. Αποχές Απορρίβεται. 288 υπέρ. Κατά. Αποχές έλεγχος. Για την 288. Die Abstimmung ist geschlossen. 56 υπέρ 11 κατά εγκρίνεται. 290 υπέρ. Κατά. Άποχες έγκρινεται. 293 υπέρ. Κατά. Άποχες έγκρινεται. 294 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 295 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 296 υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. 297 υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. 299 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 300 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 301 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 302-303 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 304 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 305 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος παρακαλώ. Πέρας. Τριακόσια υπέρ. Κατά αποχές Απορρίβεται. Έχουμε τώρα πολλές με τροπολογίες που θα συζητηθούν πολύ. 310, 11 και 12. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. 13, 313, 314 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Απορρίπτεται. 315 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Σε τμήματα ψηφοφορία για την 316-317. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Abstimmung ist geschlossen. Πέρασε. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Έναξη ψηφοφορίας. Δεύτερο τμήμα. Ψηφίζουμε. Υπέρ. Για το δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά. Απορρίπτεται. Τρίτο τμήμα, υπέρ, κατά. Αποχές, απορρίπτεται. Η 318, υπέρ, κατά. Αποχές, απορρίπτεται. 319, υπέρ, κατά. Αποχές, απορρίπτεται. Η 69. Να ελέγξουμε την 319, θέλετε. Ψηφίζουμε. Γιατί σε κάποιες περιπτώσεις ε, δεν είναι σαφές αποτέλεσμα. The vote is closed. 29 to 29 υπέρ, 36 κατά, απορρίπτεται. 69 υπέρ. Κατά. Άποχες. Έλεγχος. Πέρα ψηφορίας. «28 υπέρ δεν είναι κατά απορρίπτεται. Και τώρα περνάμε στην 3, 23, 24, 25 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 3, 26 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 327-28 υπέρ. Κατά. Άποχες. Έλαχος. Πέρα εφορίας. 32 ψήφοι υπέρ, 28 κατά, εγκρίνεται. 3, 29 υπέρ. Κατά. Άποχες. Έλεγχος. Πέρας Βορειάς. Ναι, Ευτυχώ απορρίπτεται 30 υπέρ, 31 κατά, γιατί δεν έπρεπε να την ψηφίσουμε. Γιατί είχε εγκριθεί προηγούμενη. Ψηφίζουμε λοιπόν τώρα την 3.30 υπέρ. Κατά. αποχε απορρίπτεται. 3.31 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Από. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 3... δύο. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. Η 333. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Η 334. Υπέρ. Α, όχι, όχι, όχι. Έχετε εκπαιδευτεί. Η 335. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 336. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 337. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η ε, 338 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Θέλετε έλεγχο να κάνουμε. Να κανονιστεί το έλεγχο και να συντονιστεί. Πέρας ψηφορίας. 30 υπέρ, 36 κατά, απορρίπτεται. Η 3, 39 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 3, 40 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η 3, 41, 3, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 343 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 3.44 υπέρ. Κατά. Άποχες. Έλεγχος. Πέρας ψηφορίας. 29 υπέρ, 32 κατά απορρίπτεται. Τίποτα. Η 68 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 3.45 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 19 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 369 Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Και περνάμε τώρα στην συμβαστική 20 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται, αλλά ας το ελέγξουμε για καλό και για κακό. Πέρας. 35 υπέρ, 31 κατά, εγκρίνεται. 370-371 τώρα, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 372 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 373 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 374 υπέρ. Η 373 Ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά την 373, ένα ψηφορίας. πέρασε. 11 υπέρ 52 κατά. Οριακό, λέει ο πρόεδρος. Η 374 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 3.75 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 3.76 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 3.77-3.78 υπέρ. Κατά. Ας αλλάξουμε. Εγκρίνεται. Μάλλον πρώτα ολοκληρώνεται η ψηφοφορία. Α, 26 υπέρ, 34 κατά. Απορρίπτεται. 380-381 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 382 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Το τελευταίο αυτό κομμάτι, Εργης. 384 με 387, υπέρ. Κατά. Άποχες εγκρίνεται γιατί δεν συμμετείχε η μισή επιτροπή. Συμβαστική 21 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Περνάμε στην 22. Συμβαστική 22. Στην περίφημη συμβαστική 22. Σε τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Άποχες. Έγκρινεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Άποχες. Έγκρινεται. Τρίτο τμήμα υπέρ. Κατά. Άποχες. Έγκρινεται. Και περνάμε στην 411. Αν σωστά τα βλέπω τα πράγματα. Υπέρ για την 411. Κατά αποχές απορρίπτεται. Και τώρα περνάμε στην 417. Α, διαδικαστικό. Ελένη. Θα σας παρακαλούσα η τροπολογία μου με αριθμό 414 να μπει σε ψηφοφορία γιατί δεν περιλαμβάνεται στο Compromise 22 και συγκεκριμένα η πολύ, πάρα πολύ σημαντική φράση η λύση θα πρέπει να ευθυγραμμίζεται με τις αρχές και αξίες ε, που αποτελούν τα θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Also, dieses ist... Er- Μάλιστα, αυτό αποτελεί τμήμα, πρώτο, το πρώτο τμήμα της 715 που θα ψηφιστεί. Αυτό με τις αξίες και το καθεξής. Και το άλλο τμήμα είναι αντιφατικό. Από την, μάλλον ε, είναι αντίθετο με την συμβαστική 22. Γι' αυτό θα ψηφίσουμε την 415, όπου θα βρείτε το πρώτο τμήμα σε ό,τι αφορά την αναφορά στις αξίες. 415 υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. 417 υπέρ. 417 τώρα. Υπέρ της 417. Κατά. Άποχες απορρίπτεται. Και τώρα περνάμε στην τροπολογία 422. Με προφορική τροπολογία Απορρίπτεται η προφορική τροπολογία. Αυτό λέει εδώ πέρα. Α, μάλιστα. Είναι ο κατάλογος του ΕΛΙΚ. 422 λοιπόν με προφορική τροπολογία ψηφίζουμε. Έκανα ένα λάθος. 422 όπως έχει όμως, αρχική έκδοση, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και τώρα περνάμε στην... Στην 426. Υπέρ της 426. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 428 υπέρ. Ναι, μα δεν προσέχατε. Πολύ λυπάμαι, αφού το ψηφίσαμε. Μα ήταν σαφές, ήταν σαφές. 428, υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. 431. υπέρ. Μα αυτό ψηφίσαμε. Την 428 την ψηφίσαμε. Απορρίφθηκε. Απορρίφθηκε. Μα το ελέγξουμε πάλι. Ας την ελέγξουμε την 428. Abstimmung ist geschlossen. 30 υπέρ, 34 κατά. Απορρίπτεται. Σα παρακαλώ συνάδελφοι να σηκώνετε καλά τα χέρια, παρόλο που υπάρχουν πολλέ τροπολογίε, για να μπορέσουμε να βλέπουμε καλύτερα και ε, αυτό μα κοστίζει και χρόνο. 431 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 432. Έχει αλλάξει κάτι, την ψηφίζουμε. Εγκρίθηκαν 418, 322, 323, ρωτάει ο πρόεδρος. Ψηφίζουμε την 432, λοιπόν. Αφού έχουν εγκριθεί 418, 422, 423, έχουν εγκριθεί. Ψηφίζουμε 432 στο σύνολό της. Υπέρ. Κατά. Απόχες. Απορρίπτεται. 434. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 437. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έγκρινεται. 438. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 442 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 440 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 441 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 275 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η ένα, Υπέρ. Κατά. Αποχές έγκρινεται. Η τροπολογία 2. Τη νέα έκδοση υπέρ. Κατά. Ξαναρωτώ. Υπέρ. Κατά. Έγκρινεται. Τρία, τέσσερα και πέντε Έχουν διεκπαιρεωθεί. Η έξι υπέρ. Κατά. Αποχές έλεγχος. Πέρας ψηφορίας. 34 υπέρ, 31 κατά, εγκρίνεται. Η 11 υπέρ. Κατά. απόχε. Άλλη μια φορά για την 11 παρακαλώ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Η 12 υπέρ. Αποχές απορρίπτεται. Για 14 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται από τις συμμετοχές που είδα. Ε, μα όχι. Πρέπει να συμμετέχετε στις ε, ψηφοφορίες. Δεν συμμετείχε το μισό του ΕΛΚ. Κοιτά σαφές το αποτέλεσμα. Πολύ σαφέ. Τέσσερι φορέ σα έχω ζητήσει να συμμετέχετε και να σηκώνετε τα χέρια σα. Ή αλλιώ κάθε φορά να ελέγχουμε. 13 καταπίπτει, 15 υπέρ. Κατά. Άποχε. Απορρίπτεται. 16 υπέρ. Κατά. Άποχε. Απορρίπτεται. 17-18 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 19 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 20 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 21 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 24 υπέρ. Κατά. Άποχες εγκρίνεται. 25 υπέρ. Κατά. Άποχες εγκρίνεται. 26-27 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 28 υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. Η 30 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 23 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 37-38 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 39 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 40 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Έλεγχος. Έλεγχος για τη 40. Πέρασε. 36 πέρα, 24 κατά εγκρίνεται. Και τώρα περνάμε στην 41 υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. 42 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 24 υπέρ. Κατά. Αποχές έγκρινεται. Η 47 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 51. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία τώρα. Για το τελικό κείμενο. Έναρξη ψηφοφορίας. Die Abstimmung ist geschlossen. Η έκθεση εγκρίνεται με 45 ψήφους υπέρ, 6 ψήφους κατά 12 αποχές. Συγχαρητήρια. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια. Aber όπως και στην προηγούμενη έκθεση, να ευχαριστήσω και τους κοιότητες εισηγητές και όλους όσοι συνέβαλαν στην επίτευξη των συμβαστικών λύσεων. Και τώρα τι έχουμε να κάνουμε άλλο. What's the next part? The next part is the, the MENA report. MENA report. Is I have just, uh, you have to go to Turkey. No, is he here? Yes, Peyo is here. Where? Over there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 Vamos a ir ahora con... Πάμε στην δεύτερη εξέταση της έκθεσης ε, για την ασφάλεια στην Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή και τις προοπτικές πολιτικής σταθερότητας. Ο εισηγητής μας είναι ο κύριο Πελιό. 361 τροπολογίες κατατέθηκα συνολικά και έχετε το λόγο για 5 λεπτά κύριε εισηγητά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν στα πέντε λεπτά που μου δίνετε να ευχαριστήσω τους χειώδεις συζητητές των διαφόρων ομάδων για τη συμβολή τους. Είναι ένα θέμα στο οποίο θα προσπαθήσουμε να πετύχουμε την όσο γίνεται ευρύτερη συνένεση λόγω του ευαίσθητου και στρατηγικού χαρακτήρα αυτής της έκθεσης. Είναι μια ευκαιρία, όπως είπατε και εσείς, ε, για να δείξουμε ενότητα γιατί διχασμός θα ήταν πολύ παράξενο σε αυτό το θέμα. Ε, πολύ σημαντική ήταν η συμβολή και πολλών συναδέλφων πέρα από τους κοιόδης εισηγητέ για διάφορα ζητήματα και οι συμβολές τους ήταν πάντοτε πολύτιμες. Θα ήθελα να υποδείξω πριν να έρθουμε στις συμβιβαστικές ε, ε, <clears throat> τροπολογίες υπάρχουν 33 και καλύπτουν τα, τις μισές από τις ε, τροπολογίες που αναφέρατε και θα δούμε αν όλες αυτές θα τους βρουν όλους σύμφωνος. Ε, καταρχήν, κάναμε κάποιες προσθήκες που ζητήθηκαν και που δικαιολογούνται μία προσθήκη για την Ιεμένη, γιατί όταν ξεκινήσαμε ε, δεν βρισκόμασταν στην ίδια κατάσταση και μία επίσης σημαντική προσθήκη για την ΙΣΙΑ που ζήτησαν πολλοί συνάδελφοι και δικαίωσο τροποποιήσαμε, κατανοήσαμε και επιθυμούμε να αλλάξουμε και αυτό προήλθε από όλο στις ομάδες ένα σύστημα ε, ε, για τα ανθρώπινα δικαιώματα και να τροποποιήσουμε κάπως ε, το τρίτο τμήμα για να τονίσουμε ότι όχι μόνο στηρίζουμε τη γενική στρατηγική υπέρ της δημοκρατίας αλλά και υπέρ των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Θα ήθελα αυτό να το, το, σας το αναφέρω γιατί σε κάποια ζητήματα που παραμένουν διαφορές Ε, εγώ θέλω ακόμα να προσπαθήσω. Υπάρχουν κάποιες ακόμα διαφορές ανάμεσα σε ομάδες που δεν έχουν την ίδια προέλευση. Ε, ε, κάποια στοιχεία επιβεβαιώθηκαν. Ε, όσον αφορά την ενέργεια, τη διαφθορά που μέχρι τώρα έλειπε από την έκθεση, και άρα για ένα σωρό θέματα μπορέσαμε να διευκρινίσουμε τα όσα είχαμε να πούμε. Να επιστήσω την προσοχή σας για κάποια θέματα που είναι τα πιο δύσκολα και είναι τα πιο σημαντικά όμως. Από τη μια πλευρά πρέπει να προσέχουμε πολύ τη διατύπωσή μας για το συριακό ζήτημα και για το κατά πόσο θα συμπεριληφθεί Ε, στο ψήφισμα ο Ασάντ. Υπήρξαν ε, ε, εξελίξεις όσον αφορά τις απόψεις μας, αλλά και όσον αφορά τη στρατιωτική κατάσταση επιτόπου και τις επιχειρήσεις που γίνονται εκεί. Ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει κάποιες θέσεις, αλλά θα ήταν επικίνδυνο να αλλάξουμε τη θέση του Ευρωκοινοβουλίου τη στιγμή όπου τα στρατιωτικά και τα διπλωματικά και διπλωματικές μάλλον προσπάθειες θα πρέπει να συνδυάζονται ώστε να δείξουμε σταθερό μέτωπο απέναντι στον Ασάντ. Και γι' αυτό και ήρθα σε επαφή με όλες τις ομάδες ε, για να έχουμε μια πολύ υπεύθυνη θέση σε αυτή τη δύσκολη ε, φάση. Θα καταλάβετε βέβαια ότι σε σχέση ε, με τα όσα πιστεύαμε πριν από δύο μήνες υπήρξαν εξελίξεις στις απόψεις, όμως παρόλα αυτά δεν πρέπει να αλλάξει η θέση του Κοινοβουλίου γιατί κάτι τέτοιο θα ήταν επιβλαβές για το στόχο μας. Κάτι ακόμα που θέλουμε να είμαστε πολύ προσεκτικοί στις μεταξύ μας συζητήσεις και νομίζω ότι έτσι θα μπορέσουμε να φτάσουμε σε πλούσια οι συμβιβαστικέ είναι το θέμα του Ιράν και η παρακολούθηση των συζητήσεων για το ζήτημα της, πυρηνική της πυρηνικής δύναμης και ε, πώς θα μπορέσουμε να εγγυηθούμε την περιφερειακή σταθερότητα αντί να, δημιουργηθεί εκεί, να δημιουργηθούν εκεί νέες δυσκολίες. Πολύ λεπτή ε, το ζήτημα λοιπόν της σύνταξης αυτών των, το των θεμάτων. Κατά τρίτη το λόγο υπήρξαν ε, διαφορετικές, αρκετά διαφορετικές απόψεις ε, και που θα μπορούσαν να προκαλέσουν εντάσεις, πράγμα που κατά τη γνώμη μου είναι άχρηστο άσκοπο ανάμεσα σε μια ανάλυση που θα ήθελε η τρομοκρατία να εδράζεται περισσότερο σε οικονομικούς, κοινωνικούς και πολιτιστικούς ε, λόγους και μια άλλη επιτυχή που αφορά μόνο τα θέματα ασφάλειας. Δεν έχουμε καθόλου τίποτα να κερδίσουμε εάν βρίσκουμε αίτια τελευταία στιγμή. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ένα τρομοκρατικό κίνημα το οποίο ε, ανθεί, υπήρχε και πριν από την ΤΑΕΣ, υπάρχει αυτόνομα από τα θέματα ασφάλειας πολιτικά θέματα και υπάρχει επίσης ε, αυτό το, το, ε- υπάρχουν αίτια τα οποία είναι πολλαπλά. Ε, πρέπει εμείς να τα αντιμετωπίσουμε, αλλά πρέπει να γίνει δουλειά πάνω σε όλα αυτά. Ορισμένοι θεώρησαν ότι έπρεπε να μιλήσουν περισσότερο για τους οικονομικούς ε, και κοινωνικούς λόγους στους οποίους οφείλεται η τρομοκρατία και άλλοι οι οποίοι θέλησαν να μιλήσουν περισσότερο για τα θέματα ασφάλειας, όπως ήταν φυσιολογικό και αναμενόμενο από αυτούς. Και ε, ε, εδώ πιστεύω ότι είναι λογικό όλα να τα αναφέρουμε. Μπόρεσα να πω αυτά που είναι οι απόψεις μου και θα προσπαθήσουμε να ε, συνδυάσουμε τις απόψεις για αυτές τις παλιές ε, συγκρούσεις, ε, της μακροχρόνιες, όπως ας πούμε η Παλαιστίνη-Ισραήλ. Δεν χρειάζεται διαρκώς να επιμένουμε. Έχουμε ειδική εργασία πάνω στο θέμα του ΝΤΑΕΣ και των άλλων τρομοκρατών και τρομοκρατιών και η αναθεώρηση μιας γενικής στρατηγικής της Ένωσης σε αυτή την περιοχή που είναι πολύ ευρεία. Αυτό είναι το πνεύμα στο οποίο δουλεύουμε και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε ώστε όλοι να ε, συμφωνήσουν όσο γίνεται περισσότερο με αυτή την έκθεση. Ευχαριστούμε κύριε Πέγια. Ο κύριος Πρέντα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αντικαθιστώ την κυρία Μανέσκου που είναι σκιώδη ηγήτρια της ομάδας μας, αλλά δυστυχώς κολλείται σήμερα. Θα ήθελα να συγχαρώ πρώτα απ' όλα τον εισηγητή για το έργο του και για την προσπάθεια που έχει καταβάλει. Εκτιμούμε ιδιαίτερως το διαλλακτικό πνεύμα συνεργασίας που επέδειξε και η κυρία Μανέσκο μου ζήτησε να επισημάνω κάποια θέματα που τη χάνουν και υποστήριξη τη ομάδα. Καταρχήν, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να διευκολύνει τον περιφερειακό διάλογο με συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων μερών και ιδιαίτερω ε, τη Σαουδική Αραβία, το Ιράν και την Τουρκία. Δεύτερον, επίγει και είναι απαραίτητο να σταματήσει η χρηματοδότηση του ISIS του Ισλαμικού κράτους από όλου τους φορείς της περιοχής, εφαρμόζοντας ένα αποτελεσματικό σύστημα επιβολής κυρώσεων που θα συμφωνήσει ο Σύνδεσμος Αραβικών Κρατών. Και επίση καλό θα ήταν να αναλυθούν πρωτοβουλίες Ευρωπαϊκής Ένωσης, Θα διαβάσω αγγλικά γιατί αγγλικά τα έγραψε. Ε, να ενισχύσουμε τις, ε, την δημιουργία ικανοτήτων, να καταπολεμήσουμε τη ρεσοστοικοποίηση, τον, τον Ισλαμισμό, να ενισχύσουμε την συνεργασία, να αντιμετωπίσουμε τους παράγοντες της κρίσης και να κάνουν κτήμα του στη διαδικασία αυτή οι ενδιαφερόμενες χώρες με συμμετοχή των αραβικών κρατών, συνεργασίας του κόλπου και του αραβικού συνδέσμου και άλλες περιφερειακές ε, δομές όπως το G5 Sahel. Συμφωνώ με το πνεύμα της έκθεσης ε, και την πρόταση ε, να ενισχυθεί η ασφάλεια και η σταθερότητα, ιδιαίτερα σε χώρες όπως το Μαρόκο. Είμαι βεβαία ότι θα έχουμε αγαστή συνεργασία και να καταλήξουμε σε κάποιες συμβιβαστικές τροπολογίες. Και να προσθέσω αυτά που είπε ο εισηγητής, ότι είναι πολύ σημαντικό να βρεθεί συμβιβαστική λύση για τη διατύπωση που θα χρησιμοποιήσουμε για τη Συρία. Και μπορεί να υπάρχουν διαφορές, αλλά είμαι πεπισμένος ότι θα καταλήξουμε σε θετική συμβεστική τροπολογία, λαμβάνοντας υπόψη να είμαστε συνεπείς και με την προηλημένη μας μέχρι τώρα θέση. και καλό θα ήταν να είναι συμπαγής και σαφής η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ώστε να μην αποδυναμωθεί η διαπραγματευτική μας θέση. Ευχαριστώ. Τώρα θα μιλήσω εγώ εκπροσωπώντας την ΚΟΕ, να ευχαριστήσω και εγώ τον εισηγητή μας για το έργο του. Θα προσπαθήσουμε και εμείς ε, να είμαστε συνεργάσιμοι για να καταλήξουμε συμφωνίες όπου γίνεται και με βάση το όραμά μας και τις απόψεις μας και να βρούμε τις σωστές λύσεις στα προβλήματα με βάση την αγαστή γειτονία και με σεβασμό της κυριαρχίας των τοπικών φορέων και κρατών. Δεν θα πρέπει να έχουμε διπλά μέτρα και σταθμά για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Γι' αυτό είναι και πολύ σημαντικό το θέμα της επίλυσης της σύγκρουσης της Δυτικής Σαχάρας, που είναι η μόνη ανοιχτή όπως επισημαίνει ο ΙΕ, και επίσης το θέμα της Παλαιστίνης μια σύγκρουση που επιβαρύνει τις σχέσεις και τη γεωπολιτική κατάσταση στις γειτονικές μας χώρες. Για τη Συρία είπαμε ότι θα στηρίξουμε τον κύριο Μιστούρα ε, και φυσικά θα είμαστε ελαστικοί απέναντι σε χώρες όπως το, Ιράκ, το Ιράν και ε, να δούμε θα μπορέσουμε να συμπεριλάβουμε και την ε, Συριακή κυβέρνηση στη λύση σε ό,τι αφορά το Ισλαμικό κράτος να πιέσουμε τη Σαουδική Αραβία, την Τουρκία και άλλες χώρες να σταματήσουν επιτέλους να χρηματοδοτούν άμεσα ή έμεσα τους τρομοκράτες αυτούς. Το λόγο έχει ο κύριος Σμιθ. Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να συγχαρώ τον Βενσόν για το πολύ καλό και ανοιχτό πνεύμα συνεργασίας που έχει δείξει ε, ε, ε, κατανοώ το σχολιά σου ιδιαίτερα για τη διαφθορά που είναι σημαντικό να αναφερθεί σε αυτή την έκθεση. Όλες μας οι τροπολογίες προσπαθούν να θέσουν σε κάποιο πλαίσιο τις απειλές στην ασφάλεια που έχουμε. θέλουμε να διευρύνουμε βεβαίως ε, το θέμα να δούμε γιατί και πώς ε, έχει προκύψει αυτό το πρόβλημα. Για το ISIS συγκεκριμένα ε, προσπαθήσαμε να δούμε το θέμα στο πλαίσιο του, στη Συρία και αλλού. Όμως ίσως θα έπρεπε να μιλήσουμε για την ορολογία, να συμφωνήσουμε για το πώς θα το ονομάζουμε. Νταές, ISIS, εν να ξέρουμε τι λέμε. Ε, ίσως λοιπόν θα πρέπει αυτό να συνδυαστεί με το τι χρησιμοποιείται στο Συμβούλιο. Ε, να έχουμε τον ίδια ορολογία. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε με την τροπολογία 65 είναι να θέσουμε στο επίκεντρο την ε, βοήθειά μας προς τους λαούς μετά από την Αραβική Άνοιξη. Μετά έχουμε το θέμα της διαφθοράς. Στην 140 μιλάμε για το ρόλο της κοινωνίας των πολιτών που θα πρέπει να στηρίξουμε το διάλογο, ώστε οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, να καταλάβουν ότι τους έχουμε, έχουμε στο μυαλό μας, ότι τους σκεφτόμαστε γιατί πολύ συχνά είναι οι μεγαλύτεροι μας σύμμαχοι και πολλοί έχουν χρησιμοποιήσει και καταχραστεί ε, την αντιτρομοκρατική νομοθεσία για να καταστήλουν και τους εργαζόμενους στις ΜΚΟ. Πάντως είμαι σίγουρο ότι θα βρούμε μια καλή βάση για συνένεση. Ευχαριστώ. Ο Χαουίτ. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν να συγχαρώ το φίλο Βεσσαπεγονιό είναι πολύ σημαντική έκθεση αυτή για την Επιτροπή μας και πιστεύω ότι μας κατευθύνει προς ένα ψήφισμα όπου θα έχουμε μεγάλη υποστήριξη Πολλά εδώ θα πρέπει να επενέσουμε, ιδιαίτερα του τομεί που μιλούν για εταιρικέ σχέσει με τι ελληνικοχώρε, με τον Αραβικό Σύνδεσμο, για παράδειγμα, στήριξη για την πρόοδο στην ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή. Συμφωνώ απόλυτα ε, μαζί του όσον αφορά την θέση μας ότι δεν πρόκειται να συνεργαστούμε με τον Ασάντ. Είναι πολύ επικίνδυνο να προσπαθήσουμε να ξαναγράψουμε την ε, θέση μας, να αλλάξουμε τη θέση μας με αυτό το ψήφισμα. Συμφωνώ ότι πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στην κρίση των προσφύγων. Υπάρχουν πάρα πολλά λοιπόν σε αυτή την έκθεση και νομίζω ότι είναι πολύ αποτελεσματικός. Ε, θα δούμε πώς θα ε, μπορέσουμε να ενισχύσουμε αυτή την έκθεση, ιδιαίτερα τη σχέση ανάμεσα στον ΙΠΑ, το εκπρόσωπο και τον Υπουργό ε, Εξωτερικών του Ιράν Ίσως θα πρέπει να δούμε το ψήφισμα για την Ουκρανία για να ενισχύσουμε τη θέση της ΥΠΑ της εκπροσώπου. Έχει σωστά ζητήσει να αναμεθούν περισσότερο οι Υπουργοί Εξωτερικών. Θα πρέπει να δείξουμε τη στήριξή μας προς εκείνη και ρητά επίσης να αναφέρουμε σε σχέση με την προπαγάνδα κατά των τζιχαντιστών, να το πούμε ότι πρόκειται για καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης, ότι δεν είναι πόλεμος πολιτισμών. Αυτά τα μηνύματα δηλαδή προς τους μουσουλμάνους εντός και εκτός των συνόρων μας θα είναι σαφή. Και για την εποπτεία των συνόρων επίσης κάνει κάποιες σωστές αναφορές και αυτά θα πρέπει να τα πούμε ρητά και για τη Λιβύη και για τα Παλαιστινιακά εδάφη. Μιλά για αλληλεγγύη προς τη Συρία. Ξέρω ότι προσπαθεί να κάνει σε σχέση με αυτό, αλλά πρέπει να προσέξουμε να περάσουμε ένα κείμενο που θα αναγνωρίζει ότι η ανθρωπιστική βοήθεια θα πρέπει να δοθεί και να προσφερθεί άσχετα από την πολιτική κατάσταση. Να μην παρερμηνευθεί δηλαδή η θέση μας. Επίσης, ε, κάνατε κάποιες σωστές παρατηρήσεις για την ανάπτυξη των μηνυμάτων ε, για την αστάθεια, τη σύγκρουση. Πιστεύω πως μπορούμε να τα ενισχύσουμε αυτά. Πάντως ε, και το κείμενο για την μετανάστευση νομίζω ότι θα έρθει με κάποιες ε, τροπολογίες. Θα πρέπει να δουλέψουμε για ένα ισορροπημένο κείμενο δεδομένων των συζητήσεων που γίνονται με βάση την κρίση στην Μεσόγειο Ίσως λοιπόν θα κάνετε κάποια δική σας τροπολογία για αυτό το κείμενο. Ευχαρίστω εγώ να συνεργαστώ. Πάντως είναι σημαντικά τα όσα λέτε σε σχέση με την, την ανάσχεση της τρομοκρατίας Βλέπουμε ότι δεν μας ενδιαφέρει μόνο να αντιμετωπίσουμε αυτά τα θέματα μέσα από το δικό μας πρίσμα ως Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή να ελέγξουμε την μετανάστευση και να σταματήσουμε την τρομοκρατία, αλλά ότι ενδιαφερόμαστε ε, για αυτή την περιοχή επειδή θέλουμε να προωθήσουμε την ευημερία, την ανάπτυξη πάνω απ' όλα. Αυτό το μήνυμα είναι πολύ σημαντικό να περάσει. Είναι σημαντικό να γίνουν τροπολογίες και ε, ε, συμβιβαστικές που αυτό να το αντικατοπτρίζουν. Πάντως είναι πολύ καλή η βάση για αυτή την έκθεση που είναι τόσο σημαντική. Και δεν έχω κανένα δυστυχμό για να υποστηρίξω αυτή την έκθεση και ευχαριστώ και πάλι για τη δουλειά σου. Ευχαριστώ. Και πάλι στον εισηγητή μας ο λόγος για να ολοκληρώσουμε το θέμα. Κύριε Πεγιό, σας ακούμε. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ συνάδελφοι. Για να μην μακρηγορήσω θα έλεγα ότι οι περισσότερες ανησυχίες που εκφράσατε πρώτα ο κύριος Πρέντα και κατόπιν οι υπόλοιποι συνάδουν με το πνεύμα που θα πρέπει και κατά τη γνώμη μου να διέπει τις συμβαστικέ τροπολογίες. Όπως είπε ο κύριος Χόουιτ, το δυνατό σημείο της έκθεσης αφορά την συμπερίληψη, την ανάμειξη των περιφερειακών και τοπικών φορέων του Συμβουλίου του Κόλπου, του Αραβικού Συνδέσμου, στην ανέβρεση της λύσης και θα ενισχύσουμε αυτή τη πτυχή που θα αποτελέσει και σημαντικό άξονα της έκθεσης. Να βρούμε με συνομιλητές να τους ε, πείσουμε να αναλάβουν τις ευθύνες και να συμπεριλάβουμε όσο δυνατόν περισσότερο στις συζητήσεις. Το θέμα της χρηματοδότησης επίσης αναφέρθηκε. Δηλαδή η δυνατότητα που έχουμε και η έκκληση που απευθύνουμε για πιο σαφή παρακολούθηση και αυστηρότερο έλεγχο ε, όπως είπατε και κύριε Πρόεδρε, εκ εκείνων που μπορεί να χρηματοδοτούν την τρομοκρατία. Γιατί τα τελευταία χρόνια είχαμε, δείξαμε αρκετή επίκαιρη συγκαταβατικότητα, ακόμη και διπλά μέτρα και σταθμά στο θέμα αυτό. Για το Μαρόκο είναι περισσότερο θέμα τύπου, τυπικό. Και θα πρέπει να προσθέσουμε σχέση με αυτά που είπαμε και για την Τινησία, να ενθαρρύνουμε και να βοηθήσουμε όσους ε, συμμετέχουν σε αυτή τη συζήτηση. Ε, και η αντιπροσωπεία της Λιβύης επίσης ε, θα πρέπει να αναγνωριστεί. Και για αυτά που είπατε εσείς κύριε Πρόεδρε, επαναλαμβάνω ότι αν θέλουμε απλώς να επαναλάβουμε τις θέσεις μας για τα θέματα της Δυτικής Σαχάρας της Παλαιστίνης, και στηρίζουμε την ειρηνευτική λύση τα ψηφίσματα του ΟΗΕ, τα σύνορα του 67, τα δύο κράτη και φυσικά θα πρέπει και οι διεμπλεκόμενες πλευρές να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους. Με να σταματήσουν να προκαλούν το Ισραήλ, δεν να σταματήσουν την πολιτική του επικισμού. Όλες αυτές οι θέσεις συνάδουν και συνεχίζουν τις μέχρι τώρα λιμένες θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είμαι υπέρ. Βέβαια είδα και κάποιες τροπολογίες που απάδουν από τη γραμμή αυτή και δεν επιτρέπουν την ανέβρεση κοινή λύση. Εμείς δεν θέλουμε να κουκουλώσουμε να αποφύγουμε το θέμα. Απλώς η έκθεση αυτή δεν θέλουμε να επιμένει σε θέματα που δεν σοβαρά και δεν, που δεν, δεν τα αναφέρουμε αλλού. Θέλουμε να μείνουμε σε αυτό το θέμα και δεν να μιλούμε μόνο με τη στρατηγική. Δεν μιλούμε μόνο για τη στρατηγική ασφάλεια. Φυσικά δεν θα πρέπει να ε, αποποιούμαστε των ευθυνών μας, αλλά θα πρέπει να σας υπενθυμίσω ότι και σε προηγούμενες πολιτικές και εκθέσεις είχαμε διαφορετικές τροπολογίες. Και δεν θα πρέπει να ξεφεύγουμε από το κεντρικό θέμα της έκθεσης, ε, που δεν είναι το μέα κούλπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, σε όλη την έκθεση. Φυσικά δεν ήμασταν τέλειοι, δεν τα κάναμε όλα θετικά. Και για την διαρθρωτική παρακολούθηση των Αραβικ... της Αραβικής ε, την αξιολόγηση, αλλά θα πρέπει όλα αυτά να γίνουν με ορθολογικό τρόπο, με τρόπο που δεν θα μας διχάζει, αλλά που θα μας ενώνει. Επίσης, ε, θα προσπαθήσω να ε, καλύψω τις ανησυχίες σας και φυσικά σε πνεύμα συνεργασίας κύριε Σμιθ ήταν παρόν από την αρχή των συζητήσεων. Προσπάθησα να συμπεριλάβω τις ανησυχίες σας ό,τι αφορά τη διαφθορά. Πολύ σημαντικό θέμα για να αντιληφθούμε την όλη κατάσταση και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Σας είπα ότι συμφωνούμε σε ό,τι αφορά την διεύρυνση των αιτιών. Ζητούμενο είναι η ισορροπία, όπως σας είπα και στην αρχή δεν ε, είναι μόνο δική μας ε, αμέλεια ή κάποιες ε, κοινωνικές δυσκολίες που προκαλούν την τρομοκρατία. Είναι πολύ πιο περίπλοκα τα αίτια της τρομοκρατίας και υπάρχει μια ολόκληρη ιστορία της τρομοκρατίας που έχει αρχίσει εδώ και πολλά χρόνια. Ε, επίσης, η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών μείζων ζήτημα θα πρέπει να τη διευκολύνουμε και να ενισχύσουμε και φυσικά να λάβουμε υπόψη και το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όντας συνεπείς με τις μέχρι τώρα θέσεις μας. Θέσεις μας. Ίσως θα μπορούσαμε να αναδιατυπώσουμε την αρχή του τρίτου τμήματος και τον τίτλο, ώστε να καλύπτει περισσότερες ανησυχίες. Ο κύριος Χόουιτ πολύ σωστά και εύλογα επέμεινε στο θέμα των προσφύγων. Κεντρικό ζήτημα της μέρημνας και της ανησυχίας μας και εσείς κύριε Πρέντο το είπατε, μέσω και μάκρο πρόθεσμα το θέμα των προσφύγων δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται περιστασιακά στα κατεπήγοντα, αλλά να δούμε τις ε, δεσμεύσεις μας και τις υποχρεώσεις μας και μέσω και μάκρο πρόθεσμα. Επίσης, θα πρέπει να στηρίξουμε και τις προσπάθειες της ύπατης εκπροσώπου για πολλά και διάφορα θέματα, κυρίως την αναζήτηση της ισορροπίας μεταξύ των χωρών μελών. Γιατί σε μερικές περιπτώσεις υπήρχαν και ανεπιθύμητοι ανταγωνισμοί υπερητοί και δυσάρεστη, δυσάρεστη ανταγωνιστικότητα μεταξύ των χωρών μελών. Και φυσικά θέλουμε μια κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας που θα έχει, μια, θα έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, θα είναι μεστή και θα μας καθιστά ε, σημαντικό παίκτη παγκοσμίω. Οπότε σημαντικό το θέμα της σχέσης της ΥΠΑ της εκπροσώπου και των Υπουργών Εξωτερικών προκειμένου να χρησιμοποιήσουμε στο έπακρο τι ικανότητές μας. Κύριε Χόουιτ, ζητήσατε πιο ρητές μερικές φορές εκφράσεις και φρασιολογίες, όπως είπε ο κύριος Πρέντα, σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση της μαζικής εξόδου νέων που είναι που υποκύπτουν σε αυτή την τζιχαντιστική προπαγάνδα. Και θα δούμε πώς θα ε, αναλάβουμε δράσεις ε, σχετικά. Και επίσης ε, δεν μπορούμε να ερμηνεύουμε την ε, βούλησή μας ε, για αναζήτηση κοινή στρατηγικής ε, με τη βάση του, της σύγκρουσης των πολιτισμών. Θέλουμε εκπαιδευτικό, παιδαγωγικό, θρησκευτικό διάλογο και φυσικά ενίσχυση των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, όλων των μειονοτήτων. Αυτά είναι τα βασικά επιχειρήματα και σε καμία περίπτωση επίπεδο αντιπαράθεση και σύγκρουση πολιτισμών. Θα αναζητήσουμε φυσικά ισορροπίες και στη διατύπωση για τη Συρία, για τα αίτια της τρομοκρατίας, για τα πυρηνικά του Ιράν και έχω μεγάλη αισιοδοξία για την περαιτέρω συνεργασία. Πιστεύω ότι θα καταλήξουμε σε μια έκθεση που θα συγκεντρώσει μεγάλη πλειοψηφία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γιατί μόνο έτσι η εξωτερική μας πολιτική θα έχει βάρος. Γιατί δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο μέσα στη γενική σύγχυση και το χάος να φανεί και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διχασμένο σε τόσο κέρια ζητήματα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Πεγιό. Ε, θα ήθελα επ' ευκαιρία να καλωσορίσω την αντιπροσωπεία της Μαροκινής Βουλής που πραγματοποιεί επίσκεψη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ξέρω ότι παρακολουθείτε με ενδιαφέρον την έκθεση αυτή και φαντάζομαι θα βρήκατε ενδιαφέρουσα και τη συζήτηση. Η ψηφοφορία της έκθεσης ε, θα γίνει στις 11 Ιουνίου στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων πριν παραταθεί στην ε, Ολομέλεια. Τέλος συνεδρίασης, ραντεβού στις 26 Μαΐου στην ίδια αίθουσα. Καλό σας απόγευμα.